διαδικαστικό σημείο. Σήμερα εορτάζουμε τη Διεθνή ημέρα της οικογένειας. Μια γιορτή που ορίστηκε το 1993 από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Είναι μια ευκαιρία για να προωθήσουμε τη μεγαλύτερη ενημέρωση για τα θέματα που είναι οικονομικά, κοινωνικά και δημογραφικά και αφορούν τις οικογένειες. Η οικογένεια είναι ο βασικός πυρήνας του κοινωνικού μας ιστού. Και μαζί με το σχολείο διαδραματίζει τον θεμελιώδη ρόλο της μόρφωση των νέων μας και τη μετάδοση των θεμελιωδών αξιών στις οποίες βασίζεται η κοινή μας κληρονομιά. Το Κοινοβούλιο πάντοτε βρισκόταν στο πλευρό των οικογενειών και πάντοτε υποστηρίζαμε με πυγμή την ε, σημασία να υπάρξει μεγαλύτερη εξισορρόπηση μεταξύ οικογένεια και εργασία. Αυτή την ημέρα, λοιπόν, θέλω να υπογραμμίσω θα συνεχίσουμε να αφοσιωνόμαστε και να ε, καταβάλουμε προσπάθειες για την ε, επίταξη αυτού του στόχου. κυρία Λούγκρεν. Ο κύριος Λούγκρεν. Πρόεδρε, πρόεδρε Ταγιάννη, θα ήθελα να θέσω ένα διαδικαστικό ζήτημα σε ό,τι αφορά το άρθρο 11 για μια διαδήλωση η οποία έλαβε χώρα στις 27 Απριλίου στις Βρυξέλλες έξω από την Ολομέλεια. Μια διαδήλωση ενός ε, ε, Σουηδού συναδέλφου της κυρίας Κουκ σε ό,τι αφορά την αλληλεγγύη προς ε, τον Παλαιστίνιο τρομοκράτη Μπαλιούτη, ο οποίος έχει καταδικαστεί για τρεις τρομοκρατικές επιθέσεις. Πέντε άτομα έχουν δολοφονηθεί, μεταξύ των οποίων και μια μητέρα δύο παιδιών. Επίσης, απόπειρα δολοφονία, σε συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και συνενοχή. 33 επίσης άλλους φόνους για 33 άλλους φόνους κατηγορήθηκε για του οποίου όμως δεν καταδικάστηκε λόγω έλλειψη στοιχείων. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε διαδήλωση για επίδειξη αλληλεγγύης για καταδικασμένους τρομοκράτες. Απαιτώ κύριε Ταγιάννη ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αναλάβετε σοβαρά τις ε, ευθύνες σας και να τηλευκάνετε το ζήτημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Απευθύνομαι στους συναδέλφους της Ολομέλειας για να καταγγείλω ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και 7 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπλοκάρουν τη βοήθεια στις ευνοπαθείς περιοχές της Κεντρικής Ιταλίας. Πρόκειται για μια πρόταση που θα επιτρέπεται τη χρηματοδότηση κατά 100% την ανοικοδόμηση στις περιοχές αυτές. Θυμίζω σε όλους τους συναδέλφους ότι έχουν περάσει 7 μήνες από, αυτή την καταστροφική, ε, από τον καταστροφικό σεισμό και πολλοί πολίτες ακόμη ζουν σε σκηνές και δεν έχουν καμία προοπτική για μια φυσιολογική ζωή. Είναι η στιγμή να δείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει αλλάξει και να κάνει κάτι διαφορετικό και να επιδείξουμε την αλληλεγγύη μας. Βιαστείτε. Πρέπει να νοικοδομήσουμε άμεσα. Ο εισηγητής θα προσπιστεί τη θέση του Κοινοβουλίου με την ευκαιρία των τριμερών διαλόγων και θα ασχοληθούμε με το θέμα αυτό και θα έχουμε μια θέση πολύ ξεκάθαρη. Θα θυμίσω τα όσα είπατε στον εισηγητή αλλά νομίζω ότι γνωρίζει πολύ καλά το θέμα και θα επιληφθεί. Βεβαίω θα εγκρίνει το Κοινοβούλιο την απόφαση που έχει ήδη ψηφιστεί για το θέμα αυτό. Κάρβελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στι 14 Φεβρουαρίου, εδώ στην αίθουσα αυτή, ο κ. Παπαδάκη, ένα από του μη του Κοινοβουλίου, αναφέρθηκε στο Ισραήλ ω τρομοκρατικό κράτο. σε μια σχετική συζήτηση. Αναφέρθηκε αυτό στο Προεδρείο και ε, σας, θα σας γράψω προσωπικά κύριε Πρόεδρε για να σας ρωτήσω γιατί δεν έχει αναλυφθεί οποιαδήποτε δράση. Να είμαι πολύ σαφής ε, στο θέμα αυτό και σε άλλα παρόμοια. Δεν έχω καμία πρόθεση να πνίξω πολιτικές συζητήσεις στο συντερικό αυτό το κοινοβούλιο, αλλά για κάθε παρέμβαση στην οποία δεν υπάρχει συμφωνία ζητούνται κυρώσεις, κυρώσεις που παραβιάζουν τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κινδυνεύουμε να μεταμορφώσουμε το κοινοβούλιο σε ένα είδος λογοκριτικού οργάνου. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να πνίγω τις πολιτικές συζητήσεις. Ε, μπορούμε να συμφωνούμε ότι δεν συμφωνούμε. Αλλά εάν σε κάθε παρέμβαση ε, υπάρχει λογοκρισία κατά ενό κράτου, γίνεται επίθεση σε ένα κράτο, σε κάθε περίπτωση, εφόσον δεν υπάρχει για, ε, περίπτωση για σωματικές επιθέσεις, για πολιτικές αμφισβητήσεις, δεν μπορούμε να παρεμβαίνουμε με κυρώσεις, διότι αυτό είναι επικίνδυνο και από τη μια και από την άλλη πλευρά για οποιοδήποτε θέμα για το ότι υπόθηκαν ε, λόγια ίσως ε, απαράδεκτα ή χιδέα γιατί παραβιάζαν ε, την, τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντάξει εκεί θα μπορούσαμε να τοποθετηθούμε αλλά δεν μπορούμε να παραμβαίνουμε παντού με κυρώσεις και θα θεωρήσω ότι είναι δική μου ευθύνη να αποφασίζω αν θα απειληθούν κυρώσεις ο κύριο Χριστοφόρου Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε οφείλω να καταγγείλω κύριε πρόεδρε ότι οι δύο χώρε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η ελλάδα και η κύπρο αυτή τη στιγμή που μιλάμε υφίστανται την επιθετική και επεκτατική απειλή τη Τουρκία, η οποία παραβιάζει τόσο τα χωρικά του ύδατα όσο και τι αποκλειστικέ οικονομικέ ζώνε επιβάλλοντα και ναυτικού αποκλεισμού σε χώρε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. δεν φτάνει μόνο αυτό κύριε πρόεδρε αλλά η τουρκία προχώρησε και στι απειλέ ενάντια σε Ευρωπαϊκέ εταιρείε, όπω είναι η ένικη Total για την ανόρυξη φυσικού αερίου στην περιοχή. για μας δεν δοκιμάζονται μόνο οι δύο χώρες αυτές δοκιμάζεται η αξιοπιστία της ευρωπαϊκής ένωσης παραβιάζονται κυριαρχικά δικαιώματα όχι μόνο των χωρών αυτών αλλά και της ίδιας της ευρωπαϊκής ένωσης και θεωρώ ότι οφείλουμε να πράξουμε και να πράξετε ό,τι θα κάναμε ως ευρωπαϊκό κοινοβούλιο αλλά και ως ευρωπαϊκή ένωση εάν απειλούνται ή οποιαδήποτε άλλη χώρα από τι 27 χώρε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι δεν μπορεί μια χώρα να θεωρείται υποένταξη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι και χθε η κυρία Μογκερίνη να δέχεται τον κύριο Τσελίκ με αιτήματα από την Τουρκία και την ίδια στιγμή να προσβάλλει και να προκαλεί αρχέ και αξίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι επικίνδυνη αυτή η πρακτική τη Τουρκία, δημιουργεί κινδύνου στην Ανατολική Μεσόγειο και το σημαντικότερο και το κυριότερο προσβάλλει και προκαλεί χώρε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό τον λόγο ζητούμε την αλληλεγγύη, το σεβασμό αρχών και αξιών και τη λήψη μέτρων ενάντια σε μια χώρα που προκαλεί αστάθεια στην περιοχή, που προσβάλλει τι αρχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ταυτόχρονα ζητά βοήθεια και στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε και την έγκρισή τους από την 26η και 27η Απριλίου ε, που έχουν μοιραστεί. Υπάρχουν παρατηρήσεις. Όχι, άρα τα πρακτικά εγκρίνονται όσο έχουν. Σε ό,τι αφορά τη σύνθεση των πολιτικών ομάδων,